Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση και θα ήθελα να σας ε, ενημερώσω ότι η γραπτή δήλωση για την καταπολέμηση της ε, σκλήρινσης ε, κατά πλάκα στην Ευρώπη υπογράφηκε από, από την πλειοψηφία των βουλευτών του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 123 του κανονισμού εγκρίνεται και δημοσιεύεται στο πλαίσιο του κρατάντος κειμένου. Τα ονόματα των όσων υπογράφουν θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρώτο υπογράφοντα της γραπτής δήλωσης, τον κύριο Λούχαν. Παρακαλώ. Δεν παρίσταται εδώ, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα στα όσα σας είπα. Α, όχι, εδώ βρίσκεται. Παρακαλώ κύριε Λούγαν, έχετε το λόγο. Η γραπτή δήλωσή σας είχε τους, ε, τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών. Παρακαλώ να λάβετε θέση εν συντομία. Υπέγραψαν την γραπτή δήλωση στις 20 να πούμε ότι ζητάμε από την Κομισιόν και το Συμβούλιο να υπογράψει από κοινού μια δήλωση για την σκλήση κατά πλάκας και να προωθήσει ε, θεραπείες, ε, ευέλικτες πολιτικές. Η υιοθέτηση της δήλωσης θα υποστηρίξει την εφαρμογή ε, Εξειδικευμένη κατάρτιση για τις νοσοκόμες. Επίσης, η γραπτή δήλωση θα είναι ένα κίνητρο για να ενθαρρύνει τη συζήτηση και τη δράση μέσα στην Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο και σε, άλλους, σε άλλα θεσμικά όργανα ε, και ξεπερνάει και άλλες αρρώστιες πέρα από την σκλήση κατά πλάκας, αφορά πολλές άλλες χρόνιες παθήσεις. πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Βάσει της ημερήσιας διάταξης, η ψηφοφορία γίνεται βάσει της απροσταγμένης διαδικασίας για την έκθεση της κυρίας Σαρτόρη εν σχέση με την παράταση της συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας.